Let's start, colleagues. The point number five is report on the implementation. Ε, ας αρχίσουμε, συνάδελφοι, ε, για την οδηγία 0120 για τα ελάχιστα δικαιώματα και την προστασία των θυμάτων εγκληματικών πράξεων. Καλωσορίζω τους συναδέλφους από την Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών την κοινή εξέταση των ε, ε, εκθέσεων. Ε, ο στόχος είναι παροχή επαρκούς προστασίας στους υπήκους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί όλα και περισσότεροι ζουν και εργάζονται στην Αλοδαπή και πέφτουν θύματα εγκληματικών πράξεων σε χώρες που, των οποίων δεν είναι μόνιμοι κάτοικοι. Οι συνεισηγητές που κατέθεσαν το σχέδιο για την εφαρμογή αυτού του νομοθετήματος έκαναν μια αξιολόγηση των μέτρων που έχουν ήδη αναλάβει τα κράτη-μέλη, ούτως ώστε να αναγνωριστούν τα τοπικά δικαιώματα και υποχρεώσεις αυτών των ατόμων δυνάμει τις οδηγίες, καθώς και τα εμπόδια που υπάρχουν κατά την εφαρμογή σε εθνικό επίπεδο. Σήμερα έχουμε τη δυνατότητα να ακούσουμε τις απόψεις των, του εισηγητή και των σκιωδών εισηγητών και για τις 248 τροπολογίες που έχουν κατατεθεί για αυτή την έκθεση θα δώσω το λόγο στην ε, κυρία Χάνιβολ, στη συμπρόεδρό μου, που είναι η πρόεδρος ε, της Επιτροπής Γυναικών. Ε, κυρία Χάνιβολ, ευχαριστώ. Καλωσορίσατε. Ελπίζω να έρθουν, να καταφτάσουν και άλλοι προσεχώς. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους από την Επιτροπή Ελευθεριών για την καρποφόρα συνεργασία που είχαμε και νομίζω ότι έχουμε μια πολύ χρήσιμη και συνεργατική σχέση με τις επιτροπές. Ε, πρόκειται λοιπόν για την νομική προστασία. Αυτό, αυτή η έκθεση εγκρίθηκε από τις δύο επιτροπές τελευταία κοινή συνεδρίαση και ξέρετε ότι ε, συναποτελούν το πακέτο των θυμάτων. Έτσι ονομάζεται αυτές οι δύο οδηγίες. Ε, ο στόχος είναι να αναβαθμίσουμε την οδηγία, να την ευθυγραμμίσουμε, να την καταστήσουμε πιο αποτελεσματική, ούτως ώστε τα θύματα κλιματικών πρόξεων να έχουν την ε, δέσα προστασία παντού στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου και αν βρίσκονται. Θα δώσω το λόγο στους συνεισηγητές τώρα. Θα μας παρουσιάσουν ε, <clears throat> τις θέσεις τους για τις ε, τροπολογίες. Ε, η κυρία Χιμένας Μπεσερέλ. Ευχαριστώ. Πρώτα απ' όλα, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους βουλευτές που ε, συνέβαλαν σε αυτήν την έκθεση. Οι περισσότερες τροπολογίες είναι ε, τροπολογίες οι οποίες βοηθούν ε, στην βελτίωση της ποιότητας αυτής της εκθέσεως. Κοιτάξτε, εγώ θα ξεκινήσω μιλώντας για την οδηγία αυτή που είναι οδηγία του 12, όπως άλλωστε είπε η κυρία Χόνιμπολ, ε, αφορά την δέσμη των ε, θεμάτων και δημιουργήθηκε γιατί ε, συνειδητοποίησαμε ότι δεν υπήρχε σχετική νομοθεσία για τα θύματα. Υπήρχε μονάχα η Ευρωπαϊκή Οδηγία για τα θύματα, αλλά δεν υπήρχε καμία σημαντική απόφαση παρά μονάχα μία, η οποία μάλιστα είχε εφαρμοστεί, και υλοποιηθεί και με ελληπή τρόπο. Σε αυτή την περίπτωση οι περισσότερες ε, ε, τροπολογίες αφορούν το θέμα των θυμάτων στη διάρκεια των ποινικών διαδικασιών. Εδώ βεβαίως προσπαθούμε να διευρύνουμε διαρκώς το θέμα, αλλά ε, ξεκίνησε αφορώντας τον ρόλο των θυμάτων στα πλαίσια των ποινικών διαδικασιών. Εδώ καλύπτονται και οι περιπτώσεις ε, κατά τις οποίες τα θύματα είναι και μάρτυρες. Αυτό συμβαίνει συχνά ε, εδώ ε, ε, δεν κάνουμε νομοθεσία για τα θύματα, αλλά για να στηρίξουμε τα θύματα. Αυτό βεβαίως είναι ένα θέμα που αφορά το ποινικό δίκαιο, το οποίο όμως επικεντρώνεται κυρίως στον διαπράττοντα την βιοπραγία και όχι στο θύμα. Αυτό ήθελα να το σημειώσω. Επίσης τα θύματα θα πρέπει να ε, προστατευτούν και από μία δευτερογενή θυματοποίηση. Ε, ε, είναι πάρα πολλές οι τροπολογίες 57, 70, 71 που αφορούν το θέμα αυτό. Υπάρχουν οι 51, οι 57, 178, 228. Αυτές αναφέρονται ε, στη σημασία της σύμβασης της ε, Κωνσταντινούπολεως. Ε, δεν υπήρχε αυτό στο κείμενο του 12, αλλά εδώ γίνεται αναφορά στα ευεργετήματα τα οποία μπορούν να απορρεύσουν από την επικύρωση αυτής της ε, σύμβασης, κυρίως δε όσον αφορά την παρενόκληση. παρενόχληση. Ε, η, κυρία Βεστέρα δεν είναι εδώ, ε, που γνωρίζει πάρα πολύ καλά το θέμα. Εν πάση περιπτώσει είναι εδώ η αντικαταστρατιά της, θα τα πει αργότερα ως εκπρόσωπος της Επιτροπής ΦΑΜ. Επίσης το θύμα πρέπει να έχει εγγυημένα όλα τα δικαιώματα, αυτά τα οποία αναφέρονται ήδη στο κείμενο του 12. Ε, επίσης, Υπάρχουν κάποιες τροπολογίες ε, μέσω των οποίων ε, ετούμε, θα ετούνται κάποιοι βουλευτές ε, την προστασία θυμάτων που δεν έχουν ε, ε, τα ε, έγγραφά τους τεκτοποιημένα και σε αυτή την περίπτωση αυτά τα θύματα να προστατεύονται και να μην, αντιμετωπίζουν, να λοιπόν ποινικέ διαδικασίες λόγω του ότι παρατύπως διαμένουν στη χώρα. Είναι θύματα κυρίως τράφικινγκ κλπ. Τέλος, προστασία των ε, παιδιών και χαίρομαι γιατί η κυρία Κοράτσα Μπίλτ έχει αγωνιστεί για το θέμα αυτό στο Κοινοβούλιο. Οι τροπολογίες αυτές οι οποίες αφορούν τα παιδιά και οι οποίες αφορούν ε, και την βία κατά των γυναικών, δηλαδή όταν ε, μιλάμε για θύματα ιδιαίτερως ευάλωτα, αυτές οι τροπολογίες είναι πάρα πολύ σημαντικές. Αυτή τη στιγμή στην Ισπανία έχει ξεκινήσει μια μεγάλη διαδικασία ε, ακριβώς λόγω της επίγουσας κατάστασης που έχει προκύψει από δολοφονίες μικρών παιδιών, ανηλίκων. Επίσης, ένα πρόβλημα στα κράτη-μέλη είναι ότι ε, οι επαγγελματίες του δικαίου δεν έχουν την απαραίτητη κατάρτιση ε, έτσι ώστε να ε, αντιμετωπίσουν σωστά αυτά τα προβλήματα. Αυτό έχει προκύψει ιδιαίτερος και όσον αφορά την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης. Επομένως η κατάρτιση είναι πολύ σημαντική. Επίσης, Raising Awareness Campaign. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα το οποίο το αναφέρουμε στην οδηγία του 2012 ε, γινόταν αναφορά στην σωστή ε, εφαρμογή και τον αυτοέλεγχο. Αλλά η εφαρμογή του άρθρου 22 είναι πάρα πολύ σημαντική έτσι ώστε να ληφθούν υπόψη οι ειδικέ ανάγκες των συγκεκριμένων μεμονωμένων ατόμων. Το άρθρο 22 και η διαφορετική του ε, εφαρμογή έχει προκαλέσει πολλά προβλήματα ας πούμε για τα θύματα της τρομοκρατίας. Γι' αυτό χαίρομαι που το θέμα των θυμάτων τρομοκρατικών ενεργειών σαφώς αναφέρεται σε πολλές τροπολογίες. Έχω υποβάλει πάνω από 20 τροπολογίες που αφορούν ακριβώς το θέμα των θυμάτων τρομοκρατικών ενεργειών, διότι στα πλαίσια του, ε, της προστασίας των θυμάτων υπάρχει μεγάλο ε, κενό όσον αφορά τα θύματα αυτά. Γνωρίζουμε ότι στις τελευταίες τρομοκρατικές ενέργειες στο Παρίσι, στη Νίκαια, στις Βρυξέλλες, τα θύματα δεν ε, έλαβαν εν τέλει τον ικανοποιητικό βαθμό προστασίας έτσι όπως αναφερόταν τουλάχιστον στο νομοθέτημα του 2012. Σας καλώ λοιπόν να ε, υπερψηφίσετε τις τροπολογίες αυτές. Τον Ιανουάριο στη Λίμπε μιλήσαμε για την ελληπία προστασία των ε, θυμάτων ε, της τρομοκρατικής ενέργειας του Μαρτίου στις Βρυξέλλες. Ε, είναι, και τέτοιες αναφορές των θυμάτων είχαν φτάσει και ενώπιον του ε, Βελγικού Κοινοβουλίου ε, και εκεί κατέστη σαφές ότι τα θύματα δεν δέχθησαν την σωστή αντιμετώπιση είτε από το κράτος είτε από τις κοινωνικές υπηρεσίες είτε από τις ασφαλιστικές ε, εταιρείες. Γι' αυτό λοιπόν θεωρώ ότι τα θύματα της τρομοκρατίας είναι θύματα που έχουν δεχτεί επίθεση ως πολίτες μιας χώρας και επομένως θα πρέπει να καλυφθούν όλα τα δικαιώματά τους όπως οφείλουν να καλύπτονται και τα δικαιώματα όλων των θυμάτων. Ε, θα πρέπει ειδικά δε στις περιπτώσεις θυμάτων τρομοκρατίας να καλύπτεται και η αξιοπρέπεια ε, των ε, θυμάτων. Ε, γι' αυτό λοιπόν υπάρχει η τροπολογία 203 η οποία απαγορεύει, η οποία έχει ως στόχο την απαγόρευση οποιασδήποτε θετικής αντιμετώπισης του αφηγήματος της τρομοκρατίας και ε, οπωσδήποτε την προστασία όλων των θυμάτων των τρομοκρατικών ενεργειών. Ευχαριστώ πολύ τους σκιώδεις ε, για την καλή συνεργασία. Έχουν υποβληθεί τροπολογίες οι οποίες στην πλειοψηφία τους θεωρώ ότι και σωστές είναι και αντιπροσωπεύουν ε, την κοινή γνώμη και νομίζω ότι εδώ πρέπει να ξεπεράσουμε τα κομματικά στεγανά και να αναφερθούμε στα θύματα σαν τέτοια. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ την κυρία Χιμένη. Θα δώσω τώρα το λόγο στην... Θα έδινα το λόγο στην κυρία Μλίνερ. Η Μπεατρίς ε, θα διαβάσει τα σχόλια της κυρίας Μλίνερ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Εκ μέρους λοιπόν της ε, συνεισηγήτριας ε, Αγγέλικα Μλίναρ, όπως είπε και η κυρία Χιμένεθ ήδη είπε, και εμείς από πλευρά Σάλντε χαιρετίζουμε την πολύ θετική και συνενετική συνεισφορά των συναδέλφων. Δεν βλέπουμε τροπολογίες που δεν θα μπορούσαμε να υποστηρίξουμε. Οι τροπολογίες βελτιώνουν το σχέδιο εκθέσεως είμαστε σίγουροι ότι θα έχουμε μια πλήρη και συνολική έκθεση για την προστασία των δικαιωμάτων και για την ε, σύμβαση της Κωνσταντινούπολης. Χαιρετίζουμε τις ε, τροπολογίες ε, που υπογραμμίζουν τη σημασία του μέσου αυτού για την προστασία των θυμάτων των τρομοκρατικών πράξεων. Και θα πρέπει να εξωθήσουμε αν θέλετε και τη διαδικασία επικύρωσης από πλευρά Ευρωπαϊκή Ένωσης διότι είναι ένα συνολικό και νομικά δεσμευτικό μέσο για την Ευρωπαϊκή Ένωση που βασίζεται σε τέσσερις πυλώνες αποτροπή της βίας, προστασία των θυμάτων, δίωξη και τιμωρία για τους θύτες. Δεν υπάρχει λοιπόν καλύτερο μέσο για να αντιμετωπίσουμε τη βία κατά των γυναικών και της οικογένειας, αλλά και βέβαια για να προστατεύσουμε τα θύματα. Διότι υπάρχει μια συνολική δέσμη που συμπεριλαμβάνεται για τις παραβιάσεις, για την βία μέσα στο μέσο αυτό που μας επιτρέπει να καλύψουμε πάρα πολλές επιθώς, ε, περιπτώσεις ε, σεξουαλικής εκμετάλλευσης, των παιδιών και άλλα φαινόμενα. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ και τους δύο συνεισηγητές. Ε, τα μέλη τώρα θα είχαν το λόγο, λέει η Πρόεδρος, αλλά παρακαλώ να είστε σύντομοι γιατί έχουμε χρονικές πιέσεις. Η κυρία Κοράτσα Μπίλτ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η συμπρόεδροι. Εγώ χαιρετίζω το έργο της Τερέζα και της Αγγέλικα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε μια πλήρη πολιτική προστασίας για να καταπολεμήσουμε τα φαινόμενα αυτά και να δημιουργήσουμε ένα κλίμα εμπιστοσύνης για τα θύματα παιδικής, οικογενειακής βίας, βίας κατά των, γυναικών. Πρέπει αυτά τα φαινόμενα να τα παίρνουμε σοβαρά υπόψη και εμείς και η κοινωνία συνολικά. Η έκθεση αυτή λοιπόν είναι πολύ σημαντική διότι πράγματι πρέπει να κάνουμε περισσότερα πράγματα και πιο γρήγορα ώστε να υλοποιήσουμε αποτελεσματικά την οδηγία γιατί μετά από δύο χρόνια δεν έχει μετεγγραφεί οδηγία από όλα τα κράτη-μέλη και ακόμα και αυτά που την έχουν μετεγγράψει την υλοποιούν μερικώς. Θα ήθελα λοιπόν ιδιαίτερα για ευάλωτε ομάδες όπως τα παιδιά να υπογραμμίσω τη σημασία της έκθεση αυτής και ευχαριστώ όλους του συναδέλφους που συνυπέγραψαν τροπολογίες μαζί μας για την προστασία των παιδιών ιδιαίτερα για την ενοχοποίηση, τη θυματοποίηση. Υποστηρίζω απόλυτα την ε, αρχή της πρόσβασης στη δικαιοσύνη για όλους, για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων, την αντιμετώπιση των διασυνοριακών εγκληματικών πράξεων, γιατί περί αυτού πρόκειται, τη μη διάκριση μεταξύ των θυμάτων και όπως η Τερέζα αναφέρθηκε στο άρθρο 22, αυτή η προσέγγιση που εστιάζεται στον άνθρωπο, στην προσωπικότητα, διότι δεν είναι όλοι οι ίδιοι, δεν έχουν όλοι τις ίδιες ανάγκες. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τους συναδέλφους που συνυπέγραψαν τις Προτάσει τροπολογία, Νομίζω ότι πρέπει να ενισχύσουμε ιδιαίτερα το τμήμα που αφορά στη θυματοποίηση των παιδιών. Αναφερθήκατε στο λαθρεμπόριο και ευχαριστώ Τερέζα Μπεατρίς και Αγγέλικα που υπογραμμίζεται το συσχετισμό με τη Σύμβαση Κωνσταντινούπολη, Διότι η Σύμβαση αφορά ακριβώς στην προστασία των θυμάτων. Εμείς λοιπόν με τις τροπολογίες μας καλούμε όλα τα κράτη-μέλη να επικυρώσουν και να υλοποιήσουν, να εφαρμόσουν τη σύμβαση της Κωνσταντινούπολης είναι η μόνη διεθνής συνθήκη, σύμβαση που ασχολείται με το θέμα αυτό. Και θα πρέπει τα κράτη-μέλη να συμπεριλάβουν και το stalking, την, αν θέλετε, εγκληματική παρακολούθηση, παρακολούθηση με κακό σκοπό, διότι και από κύκλους φεμινιστικούς ακούμε συχνά ότι φτάνουμε στο σημείο αυτό διότι τα θύματα δεν έχουν ληφθεί σοβαρά υπόψη σε πρώιμο σημείο και μετά είναι πολύ αργά όταν οι αρχές αναλαμβάνουν δράση επιτέλους και αυτό καταλήγει σε θανάτους. Θα ήθελα να αποτίσω τιμή και στην Ιταλο-Αιγύπτια νεαρή που σκοτώθηκε στο Λονδίνο αυτή τη βδομάδα. Την είχαν ήδη χτυπήσει πριν από ένα χρόνο. Είχαν με πολλές προειδοποίησεις και τελικώς ε, τη σκότωσαν. Έχουμε ευθύνη, θέλω να πω συνάδελφοι. Επίσης πρέπει να έχουμε περισσότερους πόρους για τις υπηρεσίες, hotline για τα θύματα, ενημέρωση που θα πρέπει να δείτε τουλάχιστον σε μία ακόμα γλώσσα εκτός εκείνης του κράτους μέλους. Διότι ακριβώς μιλούμε για διασυνοριακά εγκλήματα. Δεν πρέπει λοιπόν να είναι ελλειπής η προστασία των θυμάτων επειδή δεν μιλούν τη γλώσσα του χειριστή. Εδώ έχουμε και το κόστος της μετάφρασης. Τα κράτη-μέλη είναι σημαντικό να αναπτύξουν τις δυνατότητες αυτές στο δυναμικό αυτό, όπως και προς την ε, υποστηρίξη των υπηρεσιών και να μην αναθέτουν εξωτερικά σε μη καπαόμικρον. Η κοινωνία των πολιτών εξαιρετικό έργο κάνει, αλλά δεν αρκούν αυτά. Χρειάζεται ψυχολογική υποστήριξη μεταξύ άλλων, κοινωνικές υπηρεσίες, αποτελεσματική πρόσβαση σε όλα αυτά. Ήθελα λοιπόν να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους, τις συνεισηγήτριες και προσβλέπω με ενδιαφέρον στη συνέχιση των εργασιών μας. Σας ευχαριστώ κυρία Κάφμαν, έχει λόγο. Ευχαριστώ. Θα ήθελα καρδίως να ευχαριστήσω τις συνεισηγήτριες. Είναι εξαιρετικό το σχέδιο έκθεσης που κατέθεσαν εξαιρετικά σημαντικό και το θέμα της προστασίας των θυμάτων. Και πάντοτε ασχολούμαστε με τους δράστες, όπως σωστά είπατε, αλλά δεν ασχολείται κανείς με τα δικαιώματα των θυμάτων, δυστυχώς. Είναι καλό λοιπόν που ασχολούμαστε με αυτό, με τι κατευθυντήριε σε γραμμέ τη προστασία για να δούμε πώ εφαρμόζονται αυτέ ε, στα κράτη-μέλη. <clears throat> Κάτι άλλο σημαντικό που είπε και η κυρία Κοράτσα Μπίλτ και το οποίο κρίνω εγώ απαράδεκτο σε διάφορα κράτη-μέλη Ακόμη δεν έχουν εφαρμοστεί αυτές οι κατευθυντηρίες γραφές και αναρωτιέμαι η Επιτροπή γιατί δεν έχει υποβάλει καμία έκθεση για τη μη εφαρμογή των κατευθυντηρίων γραμμών σε αυτά τα κράτη-μέλη. Για ε, τον Νοέμβριο, από τον Νοέμβρη πέρσι θα έπρεπε να το είχε κάνει αυτό και από ό,τι φαίνεται δεν ε, θεωρεί η Επιτροπή ούτε και κάποια κρατημέλη ότι στα προτεραιότητα αυτό το θέμα. Ε, και πιστεύω ότι, ε, εγώ πιστεύω αντίθετα ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να εξετάσουμε την κατάσταση από την οπτική γωνία των θυμάτων. Θα ήθελα τώρα να σχολιάσω ένα θέμα που σχετίζεται και με τι τροπολογίε που κατέθεσα συγκεκριμένα ε, όσοι έχουν ε, καθεστώς μετανάστη. <clears throat> Τα θύματα που έχουν καθεστώ μετανάστη. Βάσει των μελετών βλέπουμε ότι ε, όσοι έχουν καθεστώς μετανάστη έχουν και υψηλότερες ε, ε, πιθανότητες να πέσουν θύματα εγκληματικών πράξεων. Επίσης φοβούνται να καταγγείλουν τη βιοπραγία και τις αξιόπινες πράξεις στην αστυνομία, διότι, παραδείγματος χάρη, φοβούνται ότι θα τους διώξουν άμα εμφανιστούν στην αστυνομία. Ε, λοιπόν, θα πρέπει να μεριμνήσουμε ότως ώστε να υπάρχουν ασφαλείς διαβλή για την καταγγελία αυτών των πράξεων ανεξαρτήτως ε, καθεστώτο, εάν πέθουν θύματα αξιόπινη πράξη να μπορούν να το καταγγείλουν και να χαίρουν της θέουσα προστασία. Θα πρέπει να προστατεύουμε από ε, την επιστροφή ε, τα, τα θύματα ε, εγκληματικών πράξεων που έχουν καθεστώς μετανάστευση. Αυτό προβλέπεται και στη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης εξάλλου. Κατά τη διάρκεια της εξέτασης της διαδικασίας θα πρέπει να προστατεύονται από, από αποπομπή και απέλαση. Ευχαριστούμε λοιπόν <clears throat> τις συνεισηγήτριες και πάλι και ας επικεντρωθούμε στην εφαρμογή των καθηγητηρίων γραμμών. Κυρία Χάνιμπολ, ευχαριστώ η κυρία Κέγκη. Eh, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και εγώ ευχαριστώ την εισηγήτρια για την εξαιρετική έκθεση, συγγήτρες για την εξαιρετική τους έκθεση. Και εγώ έχω παρουσιάσει κάποιες, υποβάλει κάποιες ε, τροπολογίες και βεβαίως και εγώ όπως και οι προηγούμενοι συνάδελφοι θα ήθελα ε, να αναφερθώ στην ιδιαίτερη προστασία των ευάλωτων ατόμων, το λέω, ε, γιατί δεν υπάρχει ακόμα σαφής ορισμός όλων των θυμάτων. Θα πρέπει να καταφέρουμε να καθορίσουμε ποια άτομα ανήκουν σε αυτήν την κατηγορία θέλουμε να καθορίσουμε στρατηγική για την αποτελεσματική προστασία όλων των θυμάτων. Αναφέρομαι κυρίως και πρώτα ε, σε, ε, ε, θέματα, σε θύματα εγκλημάτων αμίσους. Δεν μιλάμε μόνο για την κοπέλα αυτή, την Μουσταφά, η οποία δολοφονήθηκε, χτυπημένη μέχρι θανάτου, ενώ είχε ζητήσει βοήθεια. Δεν είναι μόνο αυτή, είναι και τα θύματα τα πολλά θύματα ε, τα οποία έχουν πληγεί από την ε, δολοφονική τρέλα του Λούκα Τράινη στην Ιταλία. Ακόμα ζητούν δικαίωση τα θύματα αυτά και μάλιστα μία από τις ε, ε, μάρτυρες ήταν μία γυναίκα η οποία φοβόταν, ήταν στην κατηγορία των τον άσυλο και τα φοβόταν ακόμα και για την ζωή της. Αναφερόμαστε επίσης και στα θύματα κυρίως γυναίκες του stalking της αιμονικής παραγωγής παρακολούθησης ε, γιατί αυτά τα θύματα της αιμονικής παρακολούθησης του στόκινγκ δεν αναγνωρίζονται ως θύματα σε όλες τις ε, περιπτώσεις επίσης ε, πρέπει να πούμε ότι είναι διαστηνοριακό το έγκλημα αυτό κατά των ευαλώτων θυμάτων και επομένως δεν υπάρχουν σύνορα σε αυτό θα πρέπει να δοθεί βοήθεια και αρρωγή σε όλα τα θύματα. Ευχαριστώ. Η κυρία Βερζιά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είναι πολλά τα θύματα σε όλη την ε, ε, Ευρώπη ε, και ξέρουμε ότι είναι διασυνοριακό το, το θέμα. Μπορεί να είναι θύματα και βεβαίως το νομοθέτημα του 2012 προσπάθησε να αντιμετωπίσει τα προβλήματα των θυμάτων αυτών αλλά δεν τα κατάφερε όπως υπόθηκε και από προηγούμενες ομιλήτρες. Εγώ προσωπικά ε, μπορώ να υποστηρίξω αυτά που λέει η κυρία Χιμένες ε, όσον αφορά τα θύματα της τρομοκρατίας γιατί πραγματικά ε, είναι πολυπληθή στην Γαλλία τουλάχιστον τα θύματα τρομοκρατικών ενεργειών που δεν έχουν μέχρι τώρα αποζημιωθεί. Επίσης υπάρχουν αυτά τα δευτερογενή κατά κάποιο τρόπο θύματα όπως ας πούμε στο Σεν Σεντενί, ε, που δεν έχουν ακόμα που να μείνουν, δεν έχουν αποζημιωθεί για τα σπίτια τους τα οποία καταστράφηκαν από τις εκρήξεις. Θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερω τη συζήτητρε για την ε, εργασία τους, γιατί είναι πραγματικά εξαιρετική ποιότητα. Ζητήματα πολύ σημαντικά έχουν υπογραμμιστεί όσον αφορά τα θύματα, ε, τα δικαιώματά τους και την ε, προσπάθεια αντιμετώπισης των προβλημάτων των θυμάτων. Κυρίως όταν μιλάμε για θύματα εγκλημάτων μίσου, όταν μιλάμε για θύματα τα οποία μπορεί να ανήκουν ανήκουν στην κοινότητα LGTB ε, ή που μπορεί να είναι παράτυποι μετανάστες κλπ. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να προστατευτούν και μέσα στα καταφύγια τους, μέσα στις ειδικέ δομές κλπ. <laughs> Eh, Κύριε ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε και ευχαριστώ πολύ τις εισηγήτριες για την έκθεσή τους. Ε, οι περισσότερες χώρες μέλη δεν έχουν υλοποιήσει πολιτικές ε, οι οποίες ε, να διασφαλίζουν ότι οι Eh, ε, να διασφαλίσουν τα δικαιώματα των παρατύπων μεταναστών ε, που δεν έχουν δηλαδή τα σωστά ε, ταξιδιωτικά έγγραφα. Εδώ θα ήθελα ιδίω να αναφερθώ στα θύματα όταν είναι γυναίκες και μικρά παιδιά γιατί είναι πάρα πολλά τα εγκλήματα τα οποία δεν κατονομάζονται ακριβώς λόγω του φόβου που συνδέεται με την δυνατότητα άδεια παραμονή ε, Επίση, ε, ε, Η Βουλγαρική Προεδρία δυστυχώς σε αυτήν την περίπτωση δεν θέλει από ό,τι φαίνεται να επικυρώσει τη σύμβαση της Κωνσταντινούπολεως και αυτό μας φαίνεται πολύ σοβαρό. πιστεύουμε ότι αυτά τα θύματα θα πρέπει να επικυρωσει τη συμβαση της Κωνσταντινούπολης και αυτο μας φαινεται πολυ σοβαρο πιστευουμε οτι αυτα τα θυματα θα πρεπει να τυχουν ιδιαιτερως Ιδιαίτερη αντιμετώπιση και θα πρέπει αυτοί που αντιμετωπίζουν ε, ε, τα θύματα εγκλημάτων ε, κατά των γυναικών και λόγω του φίλου τους να έχουν ιδιαίτερη κατάρτιση. Πιστεύουμε ότι θα πρέπει αυτή η μορφή της βίας να βρει οπωσδήποτε τη θέση της σε αυτή την έκθεση. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Θέλει η Επιτροπή να προσθέσει κάτι. Ενάστε και σύντομοι, αν έχετε την καλοσύνη. Ευχαριστούμε. Πολύ καλή. Πληρέστατη η έκθεση και ευχαριστούμε και για τη συζήτηση. Λοιπόν, ε, να σας ενημερώσω για τις προϊούσες εργασίες και τους τέσσερις το τομείς εξακολουθεί να είναι ψήστη σημασία η οδηγία, η εφαρμογή της δηλαδή, η ορθή εφαρμογή της Πρώτα ασχολούμαστε λοιπόν με την ελληπή εφαρμογή της. Το 16 δρομολογήσαμε μια διαδικασία μη κοινοποίηση κατά 16 κρατών μελών γιατί δεν είχαν κοινοποιήσει τα στοιχεία ε, που έπρεπε και ε, Ελλάδα τον Απρίλιο και τον Οκτώβριο την Ιρλανδία ε, εκδόθηκε σχετική κοινοποίηση. Στη συνέχεια, στο, στο ενδιάμεσο διάστημα μάλλον η Ιρλανδία, η Ρουμανία και η Σλοβενία μπόρεσαν να εφαρμόσουν σωστά την οδηγία και να μα κοινοποιήσουν τα ε, επιθυμητά στοιχεία. Ε, κρεμούν διάφορες διαδικασίες όμως ε, επί παραβάση κατά των 16 κρατών μελών για την μία έγκαιρη κοινοποίηση παρότι ε, έκτοτε έχουν δηλώσει ότι έχουν εφαρμόσει πλήρω την οδηγία. Γιατί κρεμούν οι διαδικασίε γιατί ε, εξετάζουμε τώρα τα κοινοποιημένα έγγραφα ποια μορφή έχουν και... Ε, μπορούμε ε, είτε να συνεχίσουμε με τη διαδικασία επί παραβάση, αν διαπιστώσουμε ελλείψεις, ή να κινήσουμε νέα διαδικασία. Αυτό γίνεται με εξωτερική ανάθεση. Η αξιολόγηση κάποιων κρατών μελών ε, θα ληφθεί κατά τη διάρκεια του 2018 και η συνολική μελέτη, όλα τα στοιχεία δηλαδή, θα τα έχουμε στη διάθεσή μας το 2019. Επίσης, ε, βλέπουμε στην πράξη πώς θα είναι εφαρμοστές ε, οι ρυθμίσεις της οδηγίας. Κάνουμε την επαλήθευση και εντοπίζουμε ελλείψεις που σωστά υποδείξατε ότι υπάρχουν ε, στις δύο συστάσεις σας. Ναι, θα δούμε παραδείγματος χάρη ο ορισμός του θύματος είναι πλήρης ή όχι. Ε, αν ε, δεν υπάρχει διακριτική μεταχείριση κατά των θυμάτων που δεν έχουν καθώ μόνιμη διαμονή, αν είναι εύληπτος τρόπος με τον οποίο περιγράφουμε ε, την προστασία κυρίως για όσους έχουν ειδικέ ανάγκες, να δούμε <clears throat> πώς συγκροτούνται οι υπηρεσίες υποστήριξη των θυμάτων, πώς λειτουργούν και πώς χρηματοδοτούνται. Ε, παρότι ε, αυτό δεν στα υποχρέωση των κρατών μελών. Όμως εμείς θέλουμε σφαιρική εικόνα της κατάστασης να έχουμε. Ε, επίσης, εκπαίδευση των επαγγελματιών στους τομείς αυτούς, ούτως ώστε με αξιοπρεπή τρόπο να μεταχειρίζονται τα θύματα. Αναλύουμε επίση τα δεδομένα και τα στατιστικά στοιχεία των κρατών μελών. Κανονικά έπρεπε να είχαμε πάρει τον Νοέμβρη το 2017 και ακόμα ε, τώρα λαμβάνουμε. Το 19 λοιπόν, όπως σας είπα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εκδώσει την έκθεση για την εφαρμογή της οδηγίας, γιατί τότε θα έχει τα στοιχεία στη διάθεσή της. Συνεχίζουμε πάντως ε, τη δουλειά μας. Ε, ε, ε, είχαμε διαβούλευση με 200 εμπειρογνώμονες για κυβερνήσεις κρατών μελών για την τονίσμα πόσο σημαντική είναι αυτό η οδηγία και επανέλαβαν τη δέσμευσή τους στα κράτη-μέλη για την ορθή εφαρμογή αυτής της οδηγίας. Διπλασιάσαμε και την χρηματοδότηση για, τα, για τις επιδοτήσεις για τα προγράμματα Justice και JPEG για την προστασία των θυμάτων όπως προβλέπεται στην ενωσιακή νομοθεσία 2,5 εκατομμύρια ευρώ για όλες τις επιδοτήσεις. Βοηθήσαμε και τα κράτη-μέλη για την αρμογή του πιο πρόσφατου και εκτιμένου για την προστασία των θυμάτων ε, για, τις, για την οδηγία δηλαδή ε, για τις τρομοκρατικές ενέργειες. Ε. Ένα εκατομμύριο ευρώ βρήκαμε για τη χρηματοδότηση για, τις, ε, ε, για τους εμπειρογνώμονες. Η κυρία Χάριμπολ ε, διακόπτη, μπορείτε να συντομεύετε γιατί έχουμε κι άλλα να κάνουμε. Ναι, ε, ολοκλήρωσα. Ε, τώρα, Τερέζα, θέλεις να ε, ε, συνοψίσεις όλα αυτά που ακούσαμε, να κάνεις κάποιες καταληκτικές. Τώρα μου δώσατε το λόγο. Ναι. Ναι, Πρόεδρε, καθότι πρέπει και να ψηφίσουμε, ε, θα είμαι σύντομη. Είμαι σίγουρη ότι θα δουλέψουμε καλά. Είναι σαφές ποια είναι η πλειοψηφία των ζητημάτων που και εγώ είχα σκεπτεί. Αυτό εδώ ε, που έχουμε μπροστά μας είναι μια οδηγία με ελάχιστα πρότυπα, όπως έλεγα και πριν, σχετικά με τις ποινικέ διαδικασίες υπάρχει άλλη οδηγία που αφορά στα θέματα μετανάστευσης, στα θέματα εμπορίας ανθρώπων, στα θέματα θυμάτων κατά των παιδιών. Εδώ μιλούμε για την ποινική διαδικασία της διώξης, αλλά πρέπει τα κράτη-μέλη τουλάχιστον να συμμορφώνονται με αυτά τα ολίγα που απαιτούνται διότι αν δεν συμμορφούνται προς τις διατάξεις αυτές δεν θα μπορέσουμε καν να ολοκληρώσουμε τις ποινικέ διαδικασίες σχετικά με τη δίωξη των αδικημάτων αυτών. Γιατί ε, ε, χρειαζόμαστε πράγματα απτά και συγκεκριμένα που να μπορούν να υλοποιηθούν μεταξύ των 28 κρατών μελών. Εξού και η υποστήριξή μου και προς την πρόταση τροπολογιών που έχετε υποβάλει, αλλά εδώ πρέπει να μην ξεχνούμε ότι μιλούμε για ένα συγκεκριμένο μέσο. Για τα θύματα που έχουν υποστεί βία στην Ισπανία, στην Ιταλία ή μετακινούνται μεταξύ των χωρών ή σε οποιαδήποτε άλλη χώρα και ζητούν προστασία. Δεν μπορούμε στην έκθεση αυτή να συμπεριλάβουμε βεβαίω τα πάντα. αλλά τουλάχιστον θα πρέπει να επιτύχουμε αυτά τα ελάχιστα πρότυπα που σας έλεγα. Ευχαριστούμε Τερέζα λέει πρόεδρος. Ευχαριστώ την κυρία Χόινμπολ για την συμπροεδρία και τους συναδέλφους ε, της άλλης επιτροπής. Θα ξεκινήσουμε τώρα την ψηφοφορία. Πριν από αυτό όμως θα ήθελα, συνάδελφοι, να σημειώσετε ότι έχουμε μια επίσκεψη 25 δικαστικών λειτουργών ε, και άλλων νομικών από την Πολωνία που διοργανώνεται από την μόνιμη αντιπροσωπεία της Κομισιόν στην Πολωνία. Ένα από τα θέματα που θα συζητηθούν στην επίσκεψη αυτή μελέτης είναι το κράτος δικαίου και οι τρέχουσες νομικές αλλαγές τροποποίησης στην Πολωνία η συνάντηση με τα μέλη της ΛΥΜΠΕ θα είναι 9 και 4 έως 11 στην ESP 5Ε3 αν ακούσαμε καλά την Πρόεδρο ASP διορθώση Επομένως, συνάδελφοι, τώρα για την ψήφο, την περασμένη εβδομάδα διένυμε η γραμματεία τα σχετικά, να θυμίσω σύντομα τη διαδικασία σύμφωνα με τον κανονισμό για την ίδρυση του Οργανισμού για τα Θεμελιώδη Δικαιώματα. Ορίζουμε, επικυρώνουμε τα μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής, 11 ανεξάρτητα μέλη, με υψηλή ειδικευσή στα θέματα θεμελιωδών δικαιωμάτων. Ε, με εντολή πέντε έτη μη ανανεώσιμη. Η φυστάμενη, η παρούσα εντολή εκπνέει στις 3 Ιουνίου. Έχει ζητηθεί από την Επιτροπή μας να εκφράσουμε προτίμηση μεταξύ των 21 υποψηφίων στη shortlist με μυστική ψήφο. Θα ψηφίσουμε κατά αλφαβητική σειρά και οι θετικοί ψηφοί θα ληφθούν υπόψη ώστε να καταρτιστεί μια, ένας κατάλογος προτίμησης. Σε περίπτωση ισοδυναμίας μεταξύ υποψηφίων θα καταταγούν ως ίση το Διοικητικό Συμβούλιο είχε ζητήσει από την Επιτροπή ΛΥΜΠΕ να μην δημοσιευθούν τα αποτελέσματα της ψήφου αυτής, μέχρι ότου το Συμβούλιο θα έχει υποβάλει τις προτάσεις για τα νέα μέλη Θα προχωρήσουμε τώρα στην ψήφο. Εάν θέλετε να υποστηρίξετε κάποιον υποψήφιο, παρακαλώ να ψηφίσετε υπέρ, ιδάλλως, είτε κατά είτε μπορείτε να απόσχετε. Μπορείτε να ψηφίσετε υπέρ συνολικά 11 υποψηφίων. Then open the vote. Άρχεται η ψηφοφορία, λέει πρόεδρος. Yeah, I, uh, the first candidate is 11 Bantekas. Uh, one moment. I... Μισό λεπτό λέει ο πρόεδρο. Άρχεται η ψηφοφορία το πρώτο, για το πρώτο μέλος, για τον πρώτο υποψήφιο, τον κύριο Μπαντέκα. No, sorry. Uh, uh-huh. Okay, Δεύτερος υποψήφιος. Ναι, παρακαλώ. Πρόεδρε, καθότι εδώ υπάρχει μια σύγχυση. Θα ψηφίσουμε ναι για αυτούς που θέλουμε να υπερψηφίσουμε, αυτούς που δεν επιθυμούμε πρέπει να καταψηφίσουμε ή να απόσχομαι. Μπορούμε σε αυτή την ψηφοφορία να ψηφίσουμε και κατά, λέει η Πρόεδρος. Α, ώστε πρέπει, λέει το μέλος, να ψηφίσουμε κατά. Do you prefer? Yes. Thank you. We, we would just not vote. Κοιτάξτε, μπορούμε απλά να απόσχομαι. Να ψηφίσουμε θετικά, δηλαδή, μόνο υπέρ των υποψηφίων που θέλουμε, που προτιμούμε. Η συμφωνία, λέει Πρόεδρος, είναι να μην ψηφίσουμε εφόσον δεν θέλουμε να υποστηρίξουμε. Τότε όμως, ε, Πρόεδρε, να ξαναρχίσουμε την ψηφοφορία. Λοιπόν, εντάξει, λέει η Πρόεδρος, θα επαναλάβουμε με τον πρώτο υποψήφιο, τον κύριο Μπαντέκα. Λίας Μπαντέκας. Παρακαλώ. Πίτερ Μπάρτλετ, δεύτερος υποψήφιος, άρχεται η ψηφοφορία. The Πέρας. Με συγχωρείτε, Πρόεδρε. Κατανόησα για την υπερψήφιση ή την αποχή Ή το να μην ψηφίζει, λέει μάλλον το μέλος, αλλά τι γίνεται με την αποχή. The only votes which are are positive. Κοιτάξτε, μετράμε μόνο τις θετικές ψήφους, τις ψήφους υπέρ. Μπορείτε να απόσχετε. Ο δεύτερος, λέει, πρόεδρος εννοεί ο τρίτος, υποψήφιος είναι ο Κίραν Μπράτλι, Άρχεται η ψηφοφορία και πέρας. Close. Okay, thank you. Uh, the next one is François. François Crépeau. Άρχεται η ψηφοφορία, παρακαλώ. I close the vote. Πέρας. Thanks. Uh, Επόμενος υποψήφιος, Τζον Ντασίλβα Λουίς. Luis. η ψηφοφορία. Πέρασε. Thank you. The next... Επόμενος υποψήφιος, Θεοδόρα Κωστακοπούλου Ο πρόεδρος αντιμετωπίζει δυσκολίε στην προφορά. Ψηφίζουμε. Πέρασε. Thank you, colleagues. Επόμενη υποψήφιο Τζοάννα Κουλέσσα. Άρχιτη ψηφοφορία. I close the vote. Τούβε Μαλόι, επόμενη υποψήφιο, άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Επόμενη υποψήφιο Βέρα Μέσιν. Άρχεται η ψηφοφορία και πέρας. Επόμενη προσήφιος, Άνια Μιέρ. Άρχεται ψηφοφορία. Και πέρας. Στο συγγνώμη λέει πρόεδρος. Πολύ νωρίς το είπα. Τέλος πάντων λέει πρόεδρος. Επόμενος υποψήφιο Φρανσέσκο Παλέρμο. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Επόμενη υποψήφιος Διάν Ρωμό. Ψηφίζουμε. Πέρας. Ευχαριστώ. Επόμενος υποψήφιος Άντρας Σάγιο. Ψηφίζουμε. Πέρας. Επόμενος υποψήφιος Μάρτιν Σάινιν. Ψηφίζουμε. Πέρας. Επόμενη, επόμενος υποψήφιος ο Νίκος Χράιβερ. Ψηφίζουμε. Πέρας. Επόμενος υποψήφιος Αχιλέας Σκόρδας. Ψηφίζουμε. Πέρασε. Επόμενη υποψήφιος Γιούλια Βάχινγκ. Ψηφίζουμε. Και πέρασε. Jens Βέντστετ Hansen, ψηφίζουμε παρακαλώ. Πέρας. Επόμενη υποσήφιος, Άννε Βαλ Σμιτ, παρακαλώ. Πέρας. Επόμενος υποψήφιος, John Wrench, παρακαλώ. Πέρας. And the last one... Και τελευταίος υποψήφιος, Σίνισα Ζρίνσακ. Παρακαλώ. Πέρας. Δεν θα ανακοινώσω αποτελέσματα της ψήφου. Θα κοινοποιηθούν εμπιστευτικά τα αποτελέσματα αυτά στο Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού. Και θα λάβουμε τις περαιτέρω πληροφορίες. Ζητώ συγγνώμη συνάδελφοι, αλλά έτσι προβλέπει η διαδικασία. Σας ευχαριστώ πάντως που ψηφίσατε. Και θα κάνουμε τώρα ένα διάλειμμα 5 λεπτών.